Μας. Εν τω μεταξύ, έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Πρώτον, συμμετοχή στο 7ο Φόρουμ για τη Συνοχή κατόπιν ετήματος των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιφερειών Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, ε, κληθήκαμε να ορίσουμε δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μεταβούν στο 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την πολιτική συνοχής οι συντονιστές αποφάσισαν να διορίσουν τον Γιάννα Όλμπριτς και την Ντανιέλ Λεγιώτη για ε, να ε, μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Συμμετοχή στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου για το φαντίν για τη χρηματοδότηση, ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά τα θέματα ασχοληθήκαμε και σήμερα το απόγευμα. Αυτή η διάσκεψη θα λάβει χώρα στο κτίριο Μπεχλεμό στι 6 Ιουνίου και με προσκάλεσαν με τη ιδιότητά μου του Προέδρου τη Επιτροπή Προϋπολογισμών να συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη για το funding, για τη χρηματοδότηση. Θα ε, μιλήσω στην, για τη βέλτιστη αξιοποίηση τη Ευρωπαϊκή απάντηση για τα καλύτερα εργαλεία ε, χρηματοδότηση. Και αν έχετε ιδέε, ευχαρίστω να μου τι στείλετε για να τι διαβιβάσω και να τι εκφράσω στη συζήτηση στο πάνελ που ε, θα συμμετάσχω στις 6 Ιουνίου και επιβεβαιώνω ότι εκπρόσωποι της, Ευρω... της Επιτροπής μας έχουν προσκληθεί από τον Επίτροπο Έτιγκερ στη... σε όλα αυτά τα ε, ε, καταπιστεύματα και στρατηγικές επιτροπές για την απόφαση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τη σχετική επιστολή συνυπογράφει ο πρόεδρο τη Επιτροπής Προπολογισμών και ο πρόεδρο τη Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και την απευθύνουμε διορθώνω στον Επίτροπο Έτιγκερ. Ο, ο κύριος Γκαρθία Θαμπάλ θα μας μιλήσει ε, για το θέμα που έχει αναλάβει ως βασικό βασικός και για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιρλανδίας και τη σχέση με τα σχετικά εργαλεία για τη στήριξη των εξωτερικών συνόρων και τις θεωρήσεις δεν υπάρχει ακόμα εισηγητής. Στους συντονιστές επιβεβαιώσαμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας ε, του 2018, άρα έχει βγει αυτό και έχει αποφασιστεί. Μιλήσαμε για τις ακροάσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προγραμματίζονται οι ακροάσεις αυτές για τις 19 Ιουνίου. Προθεσμία είναι 30 Μαΐου στο τέλος της ημέρας. Θα πρέπει να υποβάλλετε στη γραμματεία τα σχόλιά σας και να επιβεβαιώσετε τους ε, ε, εμπειρογνώμονες που έχουν προσκληθεί και ενδεχομένω να προτείνετε εσείς και άλλους εμπειρογνώμονες μέχρι τις 30 Μαΐου. Λέω λοιπόν ότι η συμφωνία, ξέχασα να πω, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας ε, περί αυτού πρόκειται, δεν έχουμε ακόμα εισηγητή. Σας ευχαριστώ, θεωρώ το καταλάβατε. Θα περάσουμε τώρα στο σκέλος της συνεδρίασής μας που συγγνώμη, που αφορά στην ψηφοφορία. για τον προϋπολογισμό του 2017. Γένς Γκάιερ. Δεν έχουμε αιτήματα μεταβιβάσεων, μεταφορών. Δεν έχω καμία αίτηση μεταφοράς, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ο κύριος Τάραντ είναι μαζί μας. Τον αντικαθιστάτε. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Σολέ αντικαθιστά τον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους του κυρίου Ταράν υπάρχουν δύο αιτήσει μεταφοράς. Η πρώτη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που ζητά ένα ποσό μεταφόρας 43.000 ευρώ για την χρηματοδότηση της απόκτησης ενός νέου συστήματος διαχείρισης μεταφράσεων και του λογισμικού και των αντίστοιχων υπηρεσιών που θα αφορά τόσο τις υπεργολαβικά ανατιθέμενες εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές μεταφράσεις. Και υπήρχε και άλλη μια μεταφορά κονδυλίων. Έχετε ερώτημα παρακαλώ. Και το δεύτερο αίτημα μεταφοράς μας το παρουσιάζετε. Ναι, η δεύτερη είναι από το ενεκτικό συνέδριο που ζητά την τροποποίηση του οργανόγραμματος του αφορά το μόνιμο προσωπικό. Θέλουν να μετατρέψουν μία θέση AST7 και μία θέση AST4 σε δύο μόνιμες θέσεις AT5. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από την πλευρά του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις, ο κύριος Μανκά. Όχι, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτές οι δύο μεταφορές μπορούν να θεωρηθούν ως εγκριθήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, έτσι δεν, υπάρχουν, έτσι δεν είναι. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Μόνικα Όλμαγερ, δεν υπάρχουν αιτήματα μεταφοράς που θέλετε να διατυπώσετε και ολοκληρώνουμε με τις ψηφοφορίες. Ε, δίνω τώρα το λόγο στο Γιάννη Γκάιερ για το σχέδιο διορθωτικού υπολογισμού υπαριθμών 2 στον προϋπολογισμό του 2017 που έχει να κάνει με την εγγραφή στον προϋπολογισμό των πλεονασμάτων του 16. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο πλεονάσμα στον προϋπολογισμό του 2016 το οποίο φτάνει τα 6,4 δις ευρώ που αποτελείται από τα εξής πόστα έχουμε μια υστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων δηλαδή είναι κονδυλία τα οποία δεν ξοδεύτηκαν έχουμε πρόστιμα και καταβολές επιτοκίων που έχουν καταβληθεί στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους πάνω από 3 δισεκατομμυρία ευρώ Έχουμε μια διόρθωση των ιδίων πόρων ύψος λίγο περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που ανάγεται κυρίως στο πρόβλημα της κατάπτωσης, της πτώσης μάλλον της ισοτιμίας της μπύρας τερτίνας... σε σύγκριση με το ευρώ. Εκεί αυτό συμπίπτει χρονικά με την αποφάση υπέρ του Brexit. Συζήτησαμε το πρόβλημα πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλα σημεία χρήματα επειδή τα κονδύλια που εμβάζονται στη Μεγάλη Βρετανία για τη χρηματοδότηση των δύο θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, των δύο οργανισμών των που βρίσκονται εκεί, που είναι ο Οργανισμός Τραπεζών και, και ο Οργανισμός Φαρμάκων. Τα εμβάσματα λοιπόν γίνονται σε ευρώ και λόγω της μετατροπής σε συνάλλαγμα Έχουμε 173 δις εκατομμυρία ευρώ. Σε παρακαλώ, Χάινερ, σταμάτα να μην γελάς, αλλιώς θα αρχίσω να γελάω και εγώ. Μετά από τον υπολογισμό της διαφόρας, έχουμε 1,3 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία λόγω της, χάσαμε λόγω της ε, πτώσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας τερνίνας. Στο ζήτημα της ελληπούς απορρόφησης, κανονικά είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο, εδώ έχουμε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό, το οποίο σχετίζεται προπάντων με την ελληπή υλοποίηση της κατηγορίας 1β, δηλαδή είναι τα, είναι τα κονδύλια για τα διαφορετικά ταμεία τα οποία δεν απορροφώνται κανονικά. Θυμίζω πως ήδη μία φορά τα μειώσαμε σε, μια, σε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό και πάλι υποχώρησαν. Δηλαδή η υστέρηση εδώ οφείλεται στις σπαρμένες προγνώσεις στα κράτη-μέλη. Θα προετοιμαστούμε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την κατάσταση στον επερχόμενο προϋπολογισμό, έτσι ώστε το Συμβούλιο βάσει της αποκτηθήσας εμπειρίας θα αμφισβητήσει τους αριθμούς. Όσον αφορά την πτώση της ισοτιμίας της λύρας, είπα όλα τα βασικά. Έχουμε ακόμα ένα πλεόνασμα 1,38 δισεκατομμυρίων, οπότε δεν αποφεύγουμε να διαπιστώσουμε πως ε, δεν το θεωρώ ιδιαίτερα δίκαιο εάν τα ποσά αυτά τώρα με τη μορφή τροποποίησης των χρηματικών ροών απέναντι στα κράτη-μέλη μεταφερθούν στους άλλους 27 και πιστεύω πως θα καταθέσω μια τροπολογία ο ίδιος η οποία θα λαμβάνει αυτό υπόψη και η οποία θα ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράψει το ποσό αυτό στον τελικό λογαριασμό για τον Brexit. Επειδή έχουμε την κατάσταση τη μη πραγματική επιστροφή του ποσού αυτού, αλλά οι ίδιοι πόροι του οποίου λαμβάνουμε από του εθνικού προπολογισμού μειώνονται. Και τώρα οφείλουμε να διαπιστώσουμε πω τα 1,3 δισεκατομμύρια πρέπει να τα καταβάλουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θέτω κάποιες απαιτήσεις στο σχέδιο εκθεσής μου, οι οποίες είναι γνωστές στον κύκλο των συναδέλφων. Πιστεύω πως το πλεόνασμα δεν θα πρέπει να επιφέρει μείωση των εισφορών των κρατών μελών, αλλά να παραμείνει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτά είναι πολύ λιγότερο από τα ποσά με τα οποία, για τα οποία μαλώνουμε στον τριμερή διάλογο με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν μία φορά αφήσουμε τα χρήματα μέσα, δεν θα είχαμε τόσε διαφωνίε στο Κοινοβούλιο αυτό, δηλαδή δεν θα περάσουμε με αυτό το Συμβούλιο, είναι σαφέ. Αλλά το επιχείρημα δεν μπορώ να το αποφύγω εντελώ. Εάν όμω έχουμε επανεισρωή των χρήματων αυτών, τότε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των κρατών μελών στο ότι κάποιες εθνικές εισφορές στα καταπιστευτικά ταμεία και στο Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένονται ποσά και πως τα χρήματα αυτά στους εθνικούς χρήματο προϋπολογισμούς μπορούν να καλύψουν κενά. Βέβαια ζητώ και κάτι άλλο το οποίο πλέον δεν συντρέχει. Είναι ότι όλοι περιμένουμε την τροπολογία επαριθμών 3, η οποία στο πλαίσιο της οποίας μας διαβεβαιώθηκαν πρόσθετα κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Νεολαία. Επί του παρόντος δεν έχω πληροφορίες για το ζήτημα, αλλά άτυπα έμαθα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως το άμεσο μέλλον, ίσως και σήμερα, πρόκειται να προσκομιστεί και πιστεύω πως στις μέρες αυτές είναι απαραίτητο να θυμίσουμε το Συμβούλιο πως πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί τη λειτουργικότητά του. Κυρίες και κύριοι, το Νοέμβριο συζητούσαμε στις 4 το πρωί για το κατά πόσον το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 μπορεί να γίνει αποδεκτό σε σύνδεση με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά τώρα βλέπουμε πως με παραπομπή στις εκλογές για την κάτω βουλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί πως δεν βρίσκεται σε θέση να συμφωνήσει, να εγκρίνει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφότου δύο φορές είχαμε επιτύχει ομοφωνία. Και δεν μπορώ παρά να το ονομάσω αυτό όπως το θεωρώ πως είναι. Είναι μια ομοιρία, μια ομοιρία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου από τη Βρετανική κυβέρνηση. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι για να αποδείξει την αθότητά τη είναι αμέσω μετά τι εκλογέ να δώσει τη συμφωνία τη. Αλλά στοιχηματίζω πω δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε πρέπει να ζητήσουμε την ευθύνη του Συμβουλίου επειδή χρειαζόμαστε συμφωνία, αλλά τουλάχιστον όχι αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη του πρέπει να παραμείνουν λειτουργικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Εισηγητά, οι παρατηρήσεις σας μας ανησυχούν κάπως για το επίπεδο των πληρωμών, γιατί είχαμε μείωση των πιστώσεων πληρωμών με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ύψους 7 δις 100 κάτι εκατομμυρίων και τελικά θα έχουμε υποεκτέλεση σε σχέση με τις προβλέψεις κατά 12 δις. Και αυτό δείχνει τη δυσχέρεια. Τα κράτη-μέλη δεν δεσμεύονται. Δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. Κύριε Ουρέλ, έχετε πληροφορίες, έχετε κάτι να μας πείτε για τα θέματα που έθεσε ο Γενικός μας εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όχι, νομίζω πως ε, ο κύριος Γκάιερ έκανε μια πολύ καλή σύνοψη ε, της, ε, του σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού. Όπως γνωρίζετε, το άρθρο 18 του Δημοσιονομικού Κανονισμού αναφέρει ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός πρέπει να αφορά μόνο το πλεόνασμα του προηγούμενου έτους. Όπως είπε και ο κύριος Κάιερ, τρία είναι τα κύρια στοιχεία σε αυτό το ιδιαίτερα υψηλό πλεόνασμα. Η η στέρηση στην απορρόφηση πιστώσεων που ανέρχεται στα τρία τέταρτα του συνολικού πλεονάσματος, ο αρνητικός αντίκτυπος περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου από τους ε, ίδιους πόρους, το οποίο όπως εξήγησε και ο κύριος Γκάιερ, οφείλεται στην υποτίμηση της Βρετανικής Λύρας μετά από το δημοψήφισμα το 2016, τον Ιούνιο, Επίσης, οι συνεισφορές των κρατών μελών βασίζονται στο εθνικό τους νόμισμα, καταβάλλονται μηνιαίως και μετά μεταφέρονται επίσης μηνιαίως σε ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην περίπτωση αυτή η Βρετανική λίρα έχασε σε αξία, ο αντίκτυπος επομένως στον προϋπολογισμό ήταν αρνητικός. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν αυτό το 1,5 δις που συζητάμε τώρα και επίσης πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν κονδύλια από προγράμματα και ταμεία που ε, άργησαν να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να αποτελέσουν πλέον ε, κομμάτι του προϋπολογισμού. Επίσης, τα 4,9 δισεκατομμύρια που ανάφερε ο κ. Γκάιρ δυστυχώς ε, είναι ένα ε, ποσό σωστό, όπως είπε και ο επίτροπο κ. Έτινγκερ στην ε, διοργανική συνάντηση για τις πληρωμές το Μάρτιο. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, αναφέρθηκαν αυτοί, οι οποίοι αφορούν σε η στην απορρόφηση πιστώσεων κάτω από το, ε, την κατηγορία 1β. Αυτό πλέον των 7,1 δις που ε, υπήρχαν στον διορθωτικό προϋπολογισμό 4. Μετά, εδώ, αφορούμε, ε, εδώ ε, μιλάμε αποκλειστικά για ειστέρηση στην απορρόφηση πιστώσεων ε, κάτω από την κατηγορία 1β, συνοχή και τα διδάγματα που έχουμε αγγλίσει, όπως είπε και ο Επίτροπος το Μάρτιο, μας έχουν οδηγήσει στην ανάληψη δράσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη και θα τα ενθαρρύνουν να εφαρμόσουν τα προγράμματα το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να καταφέρουν να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες αρχές για να, αρχίσει να, αρχίσουν να ρέουν τα κονδύλια. Επίσης, τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει για τον αριθμό πιστώσεων που θα ζητήσουμε για το 2018 είναι επίσης πολύ σημαντικά. Ο Επίτροπος Έτινιερ θα σας παρουσιάσει τα σχετικά αύριο. Και έχουμε επίσης απόλυτη επίγνωση του ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον έλεγχο για το 2017 και την παρακολούθηση της κατάστασης. Τα κράτη-μέλη θα δημοσιεύσουν τις επικαιροποιημένες προβλέψεις τους για το 2017 τον Ιούλιο και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, σημειώσει και θα αξιολογήσει ε, την κατάσταση για να δει αν χρειάζεται ανάληψη δράσης για το 2017. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο και τα κράτη-μέλη να καταφέρουν, όπως προβλέπετε, να εφαρμόσουν ε, αυτά που πρέπει. Τον Ιούλιο όμως θα γνωρίζουμε περισσότερα. Έκανα μια ερώτηση επίσης ο κύριος Αγκάιρ για το πότε θα υποβάλει πρόταση για την, η Κομισιόν για την Ανεργία των Νέων. Ε, στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3 υπάρχει μια πρόταση 500 εκατομμυρίων για το 2017 που θα διατεθεί στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ε, πέρυσι τον Νοέμβριο συμφωνήθηκε αυτό από το Συμβούλιο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Αυτό είχαμε προβλέψει, έτσι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων συμφωνιών. Κύριε Ντεπρέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ 100% με την έκθεση του κυρίου Γκάιερ. Ε, έχω όμως δύο υποσημειώσεις να κάνω και τις αναφέρει και ο κύριος Γκάιερ για τις συνεισφορές των κρατών μελών να είναι πολύ ιδιαίτερο να υπολογίζονται σε εθνικό νόμισμα και να μετατρέπονται σε ευρώ. Δηλαδή, ε, ε, η Βρετανική συνεισφορά υπολογίζεται σε λίρα και μετά γίνεται η μετατροπή και μπορεί να υπάρχει κέρδος από την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας, διαφυγών κέρδος. Ο κίνδυνος είναι ασθενής όταν υποτιμώνται τα εθνικά νομίσματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ανεξαρτήτως από την ε, αξία του εθνικού νομίσματος θα πρέπει το κράτος μέλος να ε, καταβάλει χι ευρώ. Εγώ ως διαπραγματευτής, αν ήμουν διαπραγματευτής, αυτό το στόχο θα είχα και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να επομιστούν την τιμή από την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας με την Βρετανική Στερλίνα που ε, προκύπτει από εσωτερική απόφαση των Βρετανών. Τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Brexit. Αυτό δεν με αφορά ή δεν είναι το βασικό. Το βασικό είναι να τροποποιήσουμε τη μεθοδολογία, να λέμε ότι η συνεισφορά υπολογίζεται σε ευρώ και έτσι θα αποφευθούν οι μεγάλες αποκλήσεις λόγω εσωτερικής απόφασης ενός κράτους μέλους που έχει να κάνει με το δικό του νόμισμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και συγκυριακός χαρακτήρας Εντάξει, αλλά το σημαντικό είναι ο δομικός. Υπάρχει ένα συγκυριακό σκέλος και ένα δομικό σκέλος και το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Συνεχώς μιλούμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με τις νέες νομοθετικές πράξεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε τις πιστώσεις και πάντοτε αναπόφευκτα υπάρχει καθυστέρηση, προθεσμία από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε την υποχρέωση μέχρι τη στιγμή που την πληρώνουμε. Μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί αυτό το χρονικό διάστημα στα πρώτα χρόνια μπορεί να έχουμε μια υποαξιοποίηση των πιστώσεων πληρωμών. Είναι δομικό αυτό, διαρθρωτικό. Αν έχετε άλλο παράδειγμα, μοιραστείτε το μαζί μου. Ευχαρίστω. Και από τη στιγμή λοιπόν που θα ξεπεράσουμε τη μισή περίοδο στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θα αρχίσουν να έρχονται τα τιμολόγια και θα αυξηθούν οι πιστώσεις πληρωμών και θα πρέπει να ε, ε, ε, δώσουμε λυσαλέα μάχη με το Συμβούλιο για να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις κτλ. Και ο κύριος Γκάιρ το λέει στο σημείο 5 και συμφωνώ απολύτως, εάν στο πλαίσιο της μελλοντική διαπραγμάτευση για το χρηματοδοτικό και χρηματοοικονομικό κανονισμό. Έχουμε μία ρήτρα που να λέει ότι όταν είμαστε εντό πλαισίου των ποσών που έχουν προβλεφθεί βάσει πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και όταν έχουμε πιστώσεις πληρωμών που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, να μπουν σε ένα χύψη απόθεμα αποθεματικών, να βρεθεί ένας μηχανισμός. Και έτσι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι στο τέλος προγραμματικής περίοδου να πηγαίνουμε να ζητιανεύουμε από το Συμβούλιο και τώρα να το πέσουμε γενναιόδοροι ε, δωρητές γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί όλες οι πιστώσεις πληρωμών. Είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα και πρέπει διαρθρωτική λύση να δοθεί. Δεν ζητάμε από τα κράτη-μέλη να πληρώσουν παραπάνω, γιατί αυτά τα οποία τους επιστρέφουμε σήμερα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους τα ζητήσουμε όταν θα αυξηθούν οι πιστώσεις πληρωμών. Ε, δεν είναι αυτό το κατάλληλο. Στο σημείο 5 ε, του κυρίου Γκάιερ ε, αναφέρεται κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε όταν θα προετοιμάσουμε τις διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το Βρετανικό Ινστιτούτο είπε πολλά ο κύριος Γκάιερ, συμφωνώ τους μαζί του. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριο Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Να προσθέσω ότι αυτή ήταν η πρόταση στην αναθεώρησή μας. Αυτό είχαμε κάνει. Προτείναμε να διατηρηθεί το πλεόνασμα εντό προπολογισμού. Και μα το αρνήθηκαν από τι πρώτε μέρε. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Εγώ αυτό πιστεύω και να το ξαναζητήσουμε και να το ξαναθέσουμε. Γιατί θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Ποιε είναι οι προβλέψει τη Επιτροπή για τον ΙΣΥΝ 3. Έχουμε ένα 2014, 15, 16. Άρα ποιες είναι οι προβλέψεις για τα χρήματα και για τα, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, commitments. Ε, στα τέλη του 17. Όντως, τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η εφαρμογή, αλλά έχει να κάνει και με τη μελλοντική συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Πώς θα κρατήσουμε στα αποθεματικά της πληρωμές και τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος, ε, να ρωτήσω το εγώ κάτι. Έχουμε ανάλυση αναχώρα της υποκατανάλωσης των πιστώσεων πληρωμών, γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Με δεδομένο το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο, ορισμένες χώρες βρίσκονται σε δημοσιονομική δυσχέρεια, δυσκολία αντιμετωπίζουν και μπορεί να έχουν την, ε, αν θέλετε, να μπουν στον πειρασμό να μην αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια 100%. Πολύ συχνά αναφέρεται ότι οι, ότι ευρωπαϊκές ενισχύσεις υποχρεώνουν το κράτος να αναλάβει υποχρέωση για νέες δαπάνες που δεν είχε αναλάβει στο παρελθόν. Και άρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο ή τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία είναι κινητήρια ή για αύξηση δημοσίων δαπανών τη στιγμή που η πολιτική στην Ευρώπη είναι να μην έχουμε επιπρόσθετες δαπάνες. Το 2014-2015 υπάρχουν πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, όμως τώρα είμαστε στο 2017 και το φαινόμενο εντείνεται, διευρύνεται. Υπάρχει δηλαδή κάτι πιο βαθύ εκεί μέσα. Ορισμένα κράτη παρετούνται από την ανάληψη υποχρεώσεων γιατί υπάρχει ένα διαφορικό που βαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό. Καλώς. τούτο λεχθέντον. Τον λόγο έχει ο Γενικός Συγητής για να ε, εξάγει συμπεράσματα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το διορθωτικό σχέδιο προϋπολογισμού υπαριθμών 2, παρόλο που πρόκειται για μεταφορά εσόδων, για εγγραφή εσόδων. Να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο κύριος Όλμπριχτ, πριν πάρει το λόγο ο κ. Γκάιερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Ντεπρέ. Πράγματι, θεωρητικά είναι εφικτό ε, μια χώρα να πληρώσει εθνικό νόμισμα. Όμως ο υφιστάμενος κανονισμός για τους ίδιους πόρους δεν το επιτρέπει. Άρα είναι κάτι το δυνατό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όχι για τώρα, όχι για σήμερα. Σε ό,τι αφορά την υποεκτέλεση των πληρωμών σε θέματα και σε πολιτικές συνοχής. Προφανώς. Είναι σημαντικό το πρόβλημα. Αλλά, χάρη στο γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ένα νέο εργαλείο, την, η συνολική μάζα για τις πληρωμές που υπάρχει από το 2014, χάρη σε αυτό το εργαλείο ανακτώ το ανακτούμε αυτά τα ποσά ε, για το ενοροφή των πληρωμών για τα επόμενα έτη και έτσι δημιουργούμε ένα επιπρόσθετο περιθώριο για να μπορούμε να πληρώσουμε τα ποσά που υποεκτελέστηκαν στις περασμένες χρονιές. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να ξαναπαίρνουμε άμεσα τα χρήματα για να τα εγγράφουμε στον προϋπολογισμό. Άλλο είναι αυτό, το είπε ο κ. Αλλά αυτό, το αρνείται ούτως ή άλλως το Συμβούλιο με το καλημέρα σας. Αλλά με αυτό το δεύτερο τρόπο που μόλις τώρα παρουσίασα μειώνεται η αρνητική αντίδραση γιατί τουλάχιστον θα έχουμε τις διαθέσιμες οροφές για να κάνουμε τις πληρωμές ε, κατά περίπτωση το 2019-2020. τώρα για το ερώτημα του 2020 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων commitments. Δεν ξέρουμε εάν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσουμε με το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013, γιατί γι' αυτό μιλάμε, να απελευθερωθούν οι υποχρεώσεις που είχαν αναλυφθεί για το προηγούμενο και μόλις κλείσουν αυτά τα προγράμματα θα έχουμε στοιχεία για τα ποσά. Είναι λίγο νωρίς σήμερα. Και τέλος για το ερώτημα του κυρίου Αχτουή για την ανάλυση αναχώρα της υποεκτέλεσης. Να πω ότι υπάρχει στο reporting που παραδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση στην αρχή του προϋπολογισμού. Έχουμε διάφορες γραφικές παραστάσεις και διάφορους πίνακες που δείχνουν την κατάσταση της εξέλιξης των παλαιών και των νέων προγραμμάτων αναχώρα. Υπάρχει μια κατάταξη, ranking, βλέπουμε τα ποσοστά των προγραμμάτων αναχώρα που έτσι όπως έχουν εκτελεστεί ήδη και βλέπουμε με σαφήνεια ποιες είναι οι χώρες που σημειώνουν καθυστέρηση και ποιες είναι οι χώρες που σημειώνουν προόδο ή που ακολουθούν τον ένα καλό ρυθμό. Αυτά ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Άρα τέλη Μαρτίου δημοσιεύθηκε αυτός ο πίνακας. Καλώς. Το έχει η γραμματεία. Πολύ ωραία. Κύριε Γενική Εισηγητά. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας. Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισής μου, είδα μόνο συμφωνία, υπάρχουν μερικές διαφορές στις αποχρώσεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις αναλύσεις των αιτίων για να παραμείνω στην εικόνα του Ζεράρ με το γιογιό που εκτείνεται λίγο πιο αργά αν συγκρίνουμε τις χρηματικές ροές με αυτές των περασμένων περιόδων χρηματοδότησης θα πρέπει να αναμένουμε μια έντονα αυξανόμενη καμπύλη προς το τέλος της περίοδου χρηματοδότησης αλλά δεν το είμαστε Οπότε έχουμε λόγω του κανόνα νυψιντρία 3 έχουμε μια παράταση προς το μέλλον και κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τις αρχές διαχείρισης και πιστοποίησης, έχουν δυσκολίες. Φυσικά πρέπει να εργαστούμε για την ροή των κονδυλίων, τα οποία έχουν επινοηθεί για τη χρηματοδότηση πολιτικής στα κράτη-μέλη. Και ανησυχώ πολύ για το μέλλον της πολιτικής συνοχής από το 2020 και μετά, όταν οι καταβολές χρημάτων εξελίσσονται ως έχουν, τότε θα βιώσουμε μια κατάσταση στην οποία σε κάποια από τα κράτη, τα οποία καταβάλουν περισσότερα από όσα εισπράττουν, θα προκύψει μια συζήτηση για το τι καλό έχει μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή η μη απορροή των χρημάτων, αν και μια τέτοια κατάσταση δεν συντρέχει. Και εφόσον ε, έχω την εικόνα εδώ, αυτοί που εδώ στην Επιτροπή αυτή προέρχονται από χώρε που καταβάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά που εισπράττουν, δεν έχουν μια τέτοια άποψη, αλλά μπορεί οι κυβερνήσει κάποιων κρατών μελών να το κάνουν. Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό. Γι' αυτό και θα χαιρόμουν αν οι συνάδελφοι σε αυτό το πλαίσιο με υποστήριζαν με τροπολογίε, αλλά έχουμε μόνο δύο μέρες καιρό επειδή 31η είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Bien. Merci. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γενικό Εισηγητή, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ τους αγαπητούς συναδέλφους και τις αγαπητές συναδέλφους που συμμετείχαν. Τροπολογίες κατατίθενται μέχρι τη μία ώρα το μεσημέρι της 4ης 31 Μαΐου και στην Επιτροπή μας θα ψηφιστεί το σχετικό θέμα είτε στις 19 είτε στις 20 Ιουνίου. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2017 υπαριθμών 3 είναι σε αναμονή και θα το συζητήσουμε όταν μας διαβιβάσει το περιεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να σας πω ότι είχαμε προβλέψει μία κατεξαίρεση συνεδρίαση της 28 Ιουνίου το απόγευμα και με αυτή την ευκαιρία ο Επίτροπος Έτιγκερ θα έρθει για να μας παρουσιάσει ένα έγγραφο προβληματισμού για τη χρηματοδότηση, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως θα μας διαφωτίσει για τις νέες αρμοδιότητες μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κατακυριευθεί από την φρενίτιδα της νέας ορμής. Μεγάλη στιγμή, 28 Ιουνίου, σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό. Είπα τα διάφορα. Έχετε κάποιο θέμα να θέσετε? Δεν βλέπω να έχετε κάτι να θέσετε, παρόλο που είστε πολλοί, εσείς οι βουλευτές που είστε παρόντες, παρόντες εδώ σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα. Θα αναστείλω τις συνεδριές, θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ για να συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 και 4 και θα έχουμε μια συναρπαστική στιγμή αύριο γιατί θα ψηφίσουμε το σχέδιο αναθεώρησης του χρηματοδοτικού κανονισμού και του όμνιμους. Μία ώρα και 45 λεπτά οι ψηφοφορίες προβλέπεται να διαρκέσουν. Και θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Όσοι από εσά είχατε προγραμματίσει να συμμετάσχετε σε μια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας πω ότι ελήψη πολεμιστών, ελήψη αγωνιζομένων, διαγωνιζομένων, αναβάλλεται αυτή η συνεδρίαση και γι' αυτό ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι παρόλα αυτά δεν το γνώρισαν και ήρθαν απόψε για αυτό λυπούμαστε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες και τις συνεργάτες μου για την εξαιρετική τους συνεισφορά, για την εξαιρετική τους διαθεσιμότητα και για την εξαιρετική τους εμπειρογνωμοσύνη. Και μιλώντας για εμπειρογνωμοσύνη θα ήθελα να μάθουμε περισσότερα για το σημείο μου που έχει να κάνει με το Brexit, γιατί τα στοιχεία τα έχει όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς δεν έχουμε τίποτα και αυτό είναι θλιβερό. Να ευχαριστήσω, λέει ο πρόεδρος και τους δερμηνείς, γιατί ξεπεράσαμε το ωράριο κατά 7 ε, λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ.